Και τώρα μια ανακοίνωση. Σύμφωνα με το άρθρο 216, σημείο 4, δεν έχει υποβληθεί κάποια αίτηση να υποβληθεί σε ψηφοφορία η διόρθωση των λαθών που ανακοινώθηκε χτες στις 5.30. Επομένως, η διόρθωση των λαθών θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Περνάμε τώρα στο κόλθο σημείο, την έκθεση της